Πορεία σήμερα στις 12. Επόμενο σημείο, έκθεση Λάινεν. Αναθεώρηση του έκτου προγράμματο δράση για το περιβάλλον και καθορισμό προτεραιοτήτων για το 7 πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον. Τον λόγο έχει ο κύριο Λάινεν. Τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το 7ο πρόγραμμα δράσης ε, για το περιβάλλον, το 6ο πρόγραμμα εκπνέει τον Ιούνιο και σκοπεύουμε βεβαίως να καταβάλουμε προσπάθειες για να βελτιώσουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Το 7ο πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι αντίγραφο του 6ου. Έχουμε προχωρήσει πολύ παραπέρα, οι προκλήσεις είναι ισχυρότερες, ε, χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση, μια οριζόντια προσέγγιση με όλους τους υπόλοιπους ε, τομείς πολιτικής. Έχουμε συστημικούς κινδύνους, τους αναφέρατε, την κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοπικιλότητας. Ε. Όλα αυτά είναι προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζονται με την κλασική πολιτική. Ε, καθώς ε, βεβαίως ε, αφορά και άλλους τομείς, ειδικά την πολιτική της ενέργειας, μεταφορών, γεωργίας, αλληλείας, την πολιτική της συνοχής, αλλά ιδιαίτερα την οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική. Και εδώ πέρα θέλω να δώσω ιδιαίτερο βάρος, είναι το δυσκολότερο μέρος, πώς θα πείσουμε τους υπουργού οικονομικών, πώς θα πείσουμε τους υπουργού οικονομίας, να ασχοληθούν με τα θέμα μας αυτά. Με το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο έχει γράψει εδώ πέρα 80 παραγράφους με προτάσεις, διαδικασίες για το 7ο πρόγραμμα δράσεις και εκεί πέρα ζητάμε να σταματήσουν οι επιδοτήσεις που βλάπτουν το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να ενσωματωθούν στις τιμές ε, ε, τα εξωτερικά κόστη, η αρχή ορυπαίνων πληρώνει και στη φορολόγηση χρειάζεται επίσης ε, μια διάσταση αηφορίας στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Υπάρχουν πολύ περισσότερες ιδέες ε, που έχουμε εδώ πέρα. Συνολικά το οικολογικό αποτύπωμα στην Ευρώπη είναι πολύ ψηλό. Αν και τα 7 δισεκατομμύρια του πλανήτη ζούσαν όπως ζουν οι Ευρωπαίοι, Οπότε δεν θα χρειαζόμασταν έναν πλανήτη, αλλά δύο. Και γνωρίζουμε πως ε, υπάρχουν όρια πλανητικά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πόρων. Γι' αυτό πρέπει η χρήση των πόρων να μειωθεί σε βαθμό ακραίο και άρα το πρόγραμμα αυτό πρέπει να ανοίξει την πόρτα για μια πράσινη οικονομία και να οδηγηθούμε σε αποτελεσματική χρήση των πόρων. Δίνουμε λοιπόν ιδιαίτερο βάρος στο αστικό περιβάλλον όπου ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι και εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε παραδειγματικές δράσεις για την χρήση των πόρων, την αποτελεσματική. Οι πράσινες πόλεις, αυτό είναι που πρέπει να γίνει στην Ευρώπη και υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα, βέλτιστες πρακτικές γενίκευσης. Η προστασία του περιβάλλοντος βεβαίως θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την προστασία της κοινωνίας των ανθρώπων, η ενσωμάτωση λοιπόν ε, της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και της υγείας θα πρέπει να ενσωματωθεί στο έβδομο πρόγραμμα πλάσιο για να βρει και έναν αντίκτυπο και μια αποδοχή. Και εδώ πέρα έχουμε κάποια κενά ακόμα. Η ρήπανση του αέρα είναι αρκετά υψηλή, η χορύπανση είναι τεράστια, ο θόρυβος είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει στην περιβαλλοντική πολιτική, υποτιμάται. Εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλά δηλητηριώδη χημικά στην ναι. Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε νέες προκλήσεις με τα υλικά και άλλα νέα υλικά τα οποία πρέπει να ερευνηθούν. Κυρίε και κύριοι, οι καλύτεροι νόμοι, τα καλύτερα προγράμματα δεν χρησιμεύουν εάν δεν τα εφαρμόσουμε και το έβδομο αυτό πρόγραμμα πρέπει να δει το έλλειμμα εφαρμογής και τέλος λέγω η Ευρώπη πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο πως εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια υφόρο διαχείριση αλλιώς η ανθρωπότητα δεν θα επιζήσει στον πλανήτη Γη Ευχαριστώ πολύ Σας ευχαριστώ κύριε Λάινεν Ο κύριος Επίτροπος Ευχαριστώ πρόεδρε Κύριε και κύριοι Ευχαριστώ τον κύριο Λάινεν για όσα έκανε για αυτή την έκθεση που είναι πράγματι επίκαιρη. Όπως ξέρετε η Κομισιόν ήδη ετοιμάζει το πρόγραμμα για το περιβάλλον για έγκριση πριν τα τέλη του χρόνου. Και μπορώ να σας πω ότι πολλές από τις ιδέες που αναφέρατε στην εισαγωγή σας είναι και δικές μας. Και νομίζω ότι θα συμπεριληφθούν στο επόμενο αυτό πρόγραμμα. Στο έκτο πρόγραμμα δημιουργήθηκε η νομοθεσία για όλους τους τομείς εκτός από το έδαφος και ανελήφθησαν νέες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα και την οικονομικότερη χρήση των πόρων μέχρι το 2020 ως συμβολή στρατηγική 2020. Όλα αυτά τώρα θα συνδυαστούν σε ένα συνεπές πλαίσιο που θα ξεπερνάει και το 2020 και θα θέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη λιγότερης χρήσης ε, διοξιδίου του άνθρακος παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά απαιτούν βέβαια πιο συνεπή λήψη αποφάσεων, πιο συνδυασμένη και συμπερίληψη αυτών των θεμάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις προτεραιότητες που θέσατε και εγώ είχα βάλει την ίδια προτεραιότητα εδώ όταν παρουσιάστηκα για πρώτη φορά εδώ στο Κοινοβούλιο και έκανα τις προγραμματικές μου δηλώσεις. «50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο χρειάζονται για την εφαρμογή των προτάσεων αυτών, αλλά η έλλειψη τέτοιων μέτρων ε, καθιστά το κόστος ακόμη βαρύτερο για την προστασία του περιβάλλοντος. Τον περασμένο μήνα η Κομισιόν υπέβαλε προτάσεις και ιδέες που θα συμπεριληφθούν και σε αυτό το 7ο πρόγραμμα που πρέπει να στοχεύει και στην καλύτερη προστασία της υγείας. Πρέπει να δούμε τι ακόμη χρειάζεται για την αντιμετώπιση της μόλυνσης γιατί υπάρχουν ακόμη ανησυχίες ότι μπορεί να μην τα καλύπτει όλα αυτά επαρκώς το υπάρχον πλαίσιο. Θα τα ξαναδούμε όλα αυτά βέβαια. Γίνονται συνεχώς αξιολογήσεις των προηγουμένως εγκριθισών οδηγιών για τα ύδατα και για το αστικό περιβάλλον που είναι και αυτό πολύ σημαντικό και στο 7ο πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες και από οικισμούς, αστικούς οικισμούς. Η διεθνής διάσταση του περιβαλλοντικού προβλήματος βέβαια είναι κάτι που επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για να εφαρμοστούν σωστά και οι διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έτσι ώστε να σεβαστούμε το στόχο της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στο 7ο πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο για τη μετάβαση σε οικονομία λιγότερο, με λιγότερες εκπομπές διοξιδίου και πέρα από το 2020. Μία μεταβατική δηλαδή προοδευτική μετάβαση που δεν θα κοστίσει υπερβολικά. Όπως πάντοτε, λαμβάνω υπόψη μας και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων. Πρέπει όλοι να κινητοποιηθούν σε όλους τους τομείς και να κάνουν ό,τι μπορούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τη συζήτησή σας θα την παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Ποτόσνικ. Η κυρία Ντάντσιλα για την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι η κληρονομιά για τις μελο... Μελο... Ε, για τους νεότερους. Η πολιτική περιβάλλοντος βέβαια από μόνη της δεν είναι αποτελεσματική. Πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό αποδεικνύεται και για τον τεράστιο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος. Βέβαια δεν θα πρέπει να δημιουργούνται προβλήματα από το περιβάλλον, από την, από την πολιτική περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη και στην οικονομία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να λάβουμε υπόψη μας τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Έχουμε ανάγκη από μια δραστήρια ε, ε, πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος ε, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τις οικονομικές παραμέτρους λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεργασία τη διαμεθοριακή με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι η μόλυνση δεν γνωρίζει σύνορα και θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τη φύση και τα οικοσυστήματα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ για μια ακόμη φορά τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντάντσιλα. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δύο λεπτά ο κύριος Φρανκό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Συγητά, σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας. Έχει ανάγκη από ένα μανιφέστο η Ευρωπαϊκή Ένωση, από μια κοινή προσπάθεια, από ένα όραμα κοινό πέραν του 2020 και γι' αυτό έχει νόημα να ξεκινάμε ένα έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον φέρνοντας σε συνέργεια όλα τα χρηματοδοτικά υπάρχοντα πλαίσια και κινητοποιώντας νέες πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε να δώσουμε εγγυήσεις για τη συνεκτικότητα των ε, περιβαλλοντικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών πολιτικών, γεωργία, αλληλεία, έρευνα, ανάπτυξη, υγεία, περιβάλλον, μεταφορές, περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και κοινωνικές πολιτικές. Παρά την οικονομική κρίση η οποία βασανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υποκύψουμε στην τυραννία του βαχυπρόθεσμου και θα πρέπει να πάρουμε μέτρα και στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η αδράνεια θα είναι μοιραία. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, ιδιαίτερα σε σχέση με την σωστή και αποτελεσματική χρήση των πόρων μας των φυσικών. Πρέπει λοιπόν με αποφασιστικότητα να επενδύσουμε στην βιώσιμη οικονομία και στην οικοκαινοτομία, γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη θα πρέπει να κάνουμε νέες αντιλήψεις, να προχωρήσουμε με νέες αντιλήψεις στην ανακύκλωση των προϊόντων, στην παραγωγή προϊόντων με ε, ε, συμβατό προς το περιβάλλον τρόπο. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και την περιβαλλοντική παιδαγωγία η οποία είναι απαραίτητη για τον Ευρωπαίο πολίτη. Έχουμε λοιπόν ένα προγραμματικό μέσο στη διάθεσή μας, έχουμε όμως και ένα μέσο επικοινωνίας. Το μέσο αυτό θα πρέπει να καταστήσει ε, ορατή και προβλέψιμη για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, για τους πολίτες, για τους επιχειρηματίες, για τους επενδυτές, όλες τις ε, δυνατότητες επένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία μας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι βάσανος. Ευχαριστώ κύριε Φρανκο. Έχει το λόγο η κυρία Ουλσκουγκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αυτό το πρόγραμμα δράσης σε δεκαετή βάση συνδέει το περιβάλλον και την υγεία. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ύδατα, τα χημικά προϊόντα κτλ. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εδώ. Θα πρέπει στο μέλλον να υπάρξει καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στην πολιτική περιβάλλοντος και τις επιμέρους πολιτικές εκτέλεσής της. υπάρχει ανάγκη θα έλεγα σαφής για σωστό έλεγχο και εφαρμογή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Ελπίζουμε αυτό το μελλοντικό πρόγραμμα να είναι φιλόδοξο παρά την οικονομική κρίση, κάτι το οποίο Ε, πρέπει να θεωρήσουμε το ε, περιβάλλον σαν πηγή ε, απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς. Και είναι πολλοί οι τομείς αυτοί. Ένα παράδειγμα. Αν ας πούμε είχαμε καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες θα χρειαζόμασταν λιγότερες επιδοτήσεις για τη μείωση των συνεπειών της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν μια πιο αποτελεσματική και αυστηρή πολιτική στο περιβάλλον να γεννήσει υπηρεσίες και θέσεις απασχόλησης. Το περιβάλλον δεν είναι μια πολιτική συνοδευτική, διακοσμητική των υπολείπων πολιτικών. Η πολιτική μας για το περιβάλλον είναι αυτόνομη, έχει σημασία και θα πρέπει ακριβώς να αποδείξουμε την αξία της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γερμπράντη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε προηγουμένως στο άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος που ε, έγινε την, αυτή τη βδομάδα στην Δανία και να αναφέρω στα αγγλικά δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να βγούμε από την οικονομική κρίση άμα δεν αναπτύξουμε την πράσινη οικονομία για να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον. Η πράσινη μεταβατική περίοδος θα δημιουργήσει περισσότερη αηφορία και ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να συγχαρώ τον Επίτροπο και την Δανική Προεδρία για αυτό το τόσο θετικό ε, ανακοίνωθεν γιατί εγώ τέτοια πράγματα από το Συμβούλιο δεν ήμουν συνηθισμένο να τα ακούω και δεν τα έχω ακούσει εδώ και πολύ καιρό. Εμείς μιλάμε για την βιοποικιλότητα και θα μιλήσουμε στο μέλλον στην Ολομέλεια τον επόμενο μήνα νομίζω για την διαφύλαξη των πόρων πρέπει να ορίσουμε και τις προτεραιότητες για το 2020 με δίκτες και δράσεις. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όμως και πιο μακριά, θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το 2050, να ορίσουμε ένα όραμα για την πράσινη Ευρώπη. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών για την οικονομία και για τα παιδιά μας διότι το greening και η οικονομία συμβαδίζουν. Ευχαριστώ τον εισηγητή Λάινεν για την εξαιρετική του εργασία και θα παρακαλούσα την Κομισιόν, την Παροτρίνο να προχωρήσει με τις προτάσεις της και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο με εξαιρετικές ιδέες. Ευχαριστώ. Κύριο Σάικχατ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Λάινεν για αυτήν την έκθεση για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Και εμείς οι πράσινοι υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό σχέδιο για το περιβάλλον. Πρέπει να εργαστούμε μια, για μια στρατηγική για το 2020 όπως είπε ο κύριος Γερμπράντη αλλά και για το 2050 να δούμε σε ποια Ευρώπη πρέπει να δουλέψουμε εμείς ε, πόσο πράσινη τη θέλουμε αυτή την οικονομία. Μόνο με πράσινη οικονομία μπορούμε να επιβιώσουμε. Είναι θεμελιώδες αυτό για το μέλλον αλλά και για το πρόγραμμα δράσης που πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Ε, πρέπει να τονίσουμε τη διεθνή διάσταση επίσης του προγράμματος και θα πρέπει να έρθω, θα, θα θέλω να σταθώ τώρα στην υλοποίηση του προγράμματος. Εμείς συνειδητοποιούμε κάθε φορά πόσο δύσκολη είναι η πραγματοποίηση αυτών των προγραμμάτων. δείτε τι γίνεται με τις offshore εγκαταστάσεις στη Βόρεια Θάλασσα, δείτε τι γίνεται με την καταστροφή σε χώρους του Natura 2000. Χρειάζεται λοιπόν η Κομισιόν να επιμείνει στην εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων για την ολοκλήρωση. Πράσινη οικονομία, όλοι μιλάνε για την πράσινη οικονομία. Υπάρχει όμως κάτι το θεμελιώδες. Δεν πρέπει να, να μιλάμε μόνο για το ΑΕΠ, πρέπει να απεφεύρουμε έναν ευρύτερο δίκτυ. Παρακαλώ λοιπόν ξεκινήστε αυτή τη στρατηγική, ξεπεράστε αυτό το όριο του ΑΕΠ Δείτε ποια θα είναι για το μέλλον τα ενεργειακά μας συστήματα. Για το 2030 χρειαζόμαστε νέους στόχους, όχι μόνο χαμηλό διοξίδιο του άνθρακος. Χρειαζόμαστε περισσότερο ενεργειακό χώρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ό,τι κάνουμε εμείς σήμερα στην Ευρώπη έχει επιπτώσεις και για τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει διεθνώς η πράσινη οικονομία να ξεκινήσει. Πρέπει εμείς λοιπόν να δώσουμε το καλό παράδειγμα με το Rio 20. Ευχαριστώ κύριε Εκχάου, το κύριο Πάσκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι επιπτώσεις του πολιτισμού στα οικοσυστήματα δημιουργούν ανεπανόρθωτη βλάβη προς το περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας να ε, περιορίσουμε αυτές τις ζημιές. Είναι πολύ εύλογες και απαραίτητες. Το 7ο αυτό πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο για την το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο για την ε, περιβαλλοντική πολιτική θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια της ε, ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Με βάση την τρέχουσα εμπειρία μας, στο επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, νομικές διατάξεις για θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να περιλάβουμε περιβαλλοντικούς στόχους σε όλες τις τομέακες μας πολιτικές. Να δώσουμε περισσότερη έμφαση και στη διασυνοριακή διάσταση της περιβαλλοντικής προστασίας. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε και τοπικές στρατηγικές με προσδιορισμένα χρονοδιαγράμματα και χρονικούς ορίζοντες και να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε ε, να αποτιμούμε τακτικά την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων. Πέραν τη γενική περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να έχουμε και ειδικέ ολοκληρωμένε πολιτικέ για του μεμονωμένου οργανισμού ή τι ε, περιφέρειες ή τι ε, αστικέ περιοχέ, λαμβάνοντα υπόψη τα ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Το 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να είναι πιο συγκροτημένο, πιο ακριβέ και πιο αποτελεσματικό για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την εμπειρία που αποκομίσαμε από την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πάσκα και τώρα έχουμε τους λοιπούς ομιλητές. Με τον κύριο Σνέρχαρτ για δύο λεπτά πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρέπει τα προγράμματα δράσεω για το περιβάλλον να εξυπηρετούν και αυτομολογούν όλοι μια μακροπρόθεσμη πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το περιβάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε όμω με το έκτο πρόγραμμα ότι αυτό πολύ υπολείπεται των προσδοκιών που οδήγησαν στην ε, θέσπιση του. το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν ε, με συναπόφαση προσδιορίσει το κείμενο με τις προτεραιότητες, ε, το κλίμα, τις φυσικούς πόρους, την ε, ποιότητα των τροφίμων, που όμως δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και αυτό το διαπιστώνουμε διότι πάνω απ' όλα στα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία, αλλά και επίσης διότι υπάρχουν πολλά εμπόδια ως προς την εξέλιξή της Βλέπουμε παραδείγματι στην έκθεση να αναφέρεται ότι υπάρχει πρόθεση για το 2020 μια ενδεικτική ανάπτυξη για μια πράσινη Ευρώπη, για ένα ε, φύλλο πορεία ε, για μια πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Μπα περιπτώσει δεν μπορώ να αναφέρω όλες τι λεπτομέρειες, δεν έχω αρκετό χρόνο, αλλά προγράμματα, δράσεις, στρατηγικέ, συγκεκριμένε πρωτοβουλίε θα έπρεπε να οδηγούν στην απαραίτητη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, πράγμα το οποίο δεν εξασφαλίστηκε πάντοτε. Πρέπει να θεσπιστούν νέοι δείκτε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση γραφειοκρατική, ε, δίκτες οι οποίοι θα στηρίξουν την εξέλιξη, την ανάπτυξη γενικότερα στις κοινωνίες μας και έτσι θα υλοποιηθούν αυτοί στα όχι. Διαφωνώ λοιπόν εδώ με τον εισηγητή που ε, λέει ότι θα πρέπει να έχει οριζόντια υλοποίηση το πρόγραμμα. Όχι, διαφωνώ, πρέπει να είναι τομεακή η προσέγγιση και η εφαρμογή. Διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εναρμόνιση άνωθεν χωρίς ε, προηγούμενη εξισορρόπηση των διαφορών. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μέρκης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του και θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης γιατί πράγματι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα συνολικά και μένει και στο θέμα της εφαρμογής. Ευχαριστώ και, για τον, και τον Επίτροπο, γιατί φαίνεται ότι και αυτός επιμένει στο 7ο πρόγραμμα. Το θέμα δεν είναι μόνο το περιβάλλον. Έχουμε να κάνουμε με το σύνολο των οικονομικών τομέων, μεταφορές, δημόσια υγεία, το σύνολο των τομέων που απασχολούν την κοινωνία. Το περιβάλλον λοιπόν είναι κοινωνική και οικονομική πολιτική και στο μέλλον θα είναι ακόμα περισσότερο. Δύο επιμέρους σημεία τώρα τα οποία με απασχολούν. Πάρα πολύ συχνά ασχολούμεθα με τις νέες τεχνολογίες με τις οποίες δεν έχουμε και απόλυτη βεβαιότητα για την αποτελεσματικότητά τους. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους που βάζουμε. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος σαν παράδειγμα στη βιομάζα. Είναι σαφές ότι στο μέλλον πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτού του είδους τους πόρους. Αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ βιαστικοί και ενθουσιώδεις για τη βιομάζα. Ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό και για διαφορετικούς λόγους. Κύριε Επίτροπε, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η εφαρμογή των αποφάσεων, αλλά με τη βιομάζα τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε τη βιομάζα έτσι ώστε να μειώσουμε πράγματι την εκπομπή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και θυμίζω επίσης ότι αντίστοιχα προβλήματα οριμότητας έχουμε και με τις νανοτεχνολογίες. Η κυρία Ρίς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας ξεκίνησε υπενθυμίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει να διασώζουμε ε, το περιβάλλον και να το έχουμε πάντα ε, σαν μία βασική μας προτεραιότητα. Πολλές φορές στις εθνικές πολιτικές και στα μέσα ενημέρωσης το περιβάλλον αγνοείται πλήρως και το ίδιο φαίνεται και στην γαλλική προεκλογική εκστρατεία. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι καλό και μάλιστα μπορούμε να το κάνουμε και με ευθυνό τρόπο. Τώρα στο 3, ε, σημείο 3 ε, υπάρχει μία αναφορά ε, στην παραγωγή του καπνού. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βοηθάμε σε καμία περίπτωση δραστηριότητες οι οποίες απειλούν την υγεία. Το περιβάλλον και η υγεία είναι αναπόσπαστα. Ήδη από τη δική μου έκθεση ε, το 2003 λέγω ότι θα πρέπει να μειώσουμε την έκθεση του πληθυσμού σε αυτό το απέσιο κοκτέιλ επικίνδυνων χημικών ουσιών. Έτσι θα καταπολεμήσουμε ε, και την ασθένεια του Αλτσχάιμερ και τους καρκίνους κτλ. Ευχαριστώ κύριε Ρης. Κυρία Χάση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θερμά ευχαριστώ προς τον εισηγητή μας, τον ε, Γιώ Λάινεν, για την πολύ αξιόλογη έκθεση του και το θαυμάσιο έργο του. Το έβδομο ε, πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό και είναι κρίμα που καθυστερούμε τόσο στη συζήτηση. Γιατί καθημερινά λαμβάνονται απο, αποφάσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον. Για παράδειγμα, στη γεωργική πολιτική. Η επίπτωση της γεωρικής πολιτικής είναι τεράστια και στην βιοπικιλότητα και στην ποιότητα του ύδατο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βαλτική θάλασσα. Η κοινή γεωρική πολιτική θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη Βαλτική θάλασσα, που είναι από τις πιο μολυσμένες θάλασσες στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη ρήπανση. Και τα αποτελέσματα της ε, γεωργίας εκεί είναι ολέθρια έχουμε αζωτούχε ενώσει και λοιπάσματα που περνούν από τους ποταμού προς τη θάλασσα και αν δεν περιοριστούν θα συνεχίσει η Βαλτική να είναι από τι θάλασσε με τη μεγαλύτερη ρήπανση στον κόσμο. Και θα έχουμε για χρόνια ολόκληρα ε, λίματα που θα επιπλέουν στα νερά τη Βαλτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσω γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πιστεύω ότι αυτό το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμο. Αλλά θα πρέπει να βασίζεται σε μια εικόνα για το μέλλον η οποία να δέχεται την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη και μια σαφέστατα αποτελεσματικής αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να δώσει εγγυήσει στην πιο σωστή εφαρμογή των νέων νομικών ρυθμίσεων πριν θέσουμε επιπλέον περιορισμούς και στόχους. Για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές απειλές θα πρέπει να στραφούμε στο μέλλον. Θα πρέπει όμως να έχουμε συγκεκριμένες αποδεδειγμένες μεθόδους και αναφέρομαι εγώ στο 23 το οποίο αναφέρεται στο περιβαλλοντικό ίχνος. Αυτό είναι μια εμπορική, εμπειρική εικόνα της πραγματικότητας και όχι η πραγματικότητα η ίδια. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να υπολογίσουμε έτσι όπως ζητείτε την ποιότητα του περιβάλλοντος. Έχω επιφυλάξεις λοιπόν και παρακαλώ να τις λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Καρτίνη. Ο κύριος Σπέραγιο Ροδρίγες, 1,5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία από τι πρώτε πρωτοβουλίε που ανέλαβα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω Ευρωβουλευτή είναι να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν προέβλεψε να συνεχίσει το έκτο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον. Τότε μου έλεγαν ότι με του μηχανισμού που είχαμε τότε ε, δεν χρειαζόταν να εξασφαλίσουμε μία συνέχεια. Τώρα κάπως καθυστερημένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί ένα κοινό άξονα των κοινοτικών πολιτικών, ένα κοινό περιβαλλοντικό οίκο, ένα σημείο αναφοράς για τα προγράμματα δράσης, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Ε, είδαμε στην, στην Καταλωνία κάποιες εγκαταστάσεις για την ε, ανακύκλωση των ε, ψυγείων. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε μέχρι 95%. Όλη αυτή η πολιτική ανακύκλωση και διαχείριση των λιμάτων χρήζουν συντονισμού για να φτάσουμε το 2032 σε 100% ανακύκλωση. Και αν, ανακύκλωση. Και αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020 χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Χαίρομαι που μία από τις προτάσεις προβλέπει το, συμβου... το το πρόγραμμα να συμβάλλει στη διαχείριση των λιμάτων και θα πρέπει να καταγγείλουμε τις ε, κυβερνήσεις που με πρόσχημα την κρίση και τη λιτότητα ε, περικόπτουν τις ε, ερευνητικέ προσπάθειες ε, και τα προγράμματα διαχείριση λιμάτων που υποθηκεύονται ουσιαστικά το μέλλον της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει η κρίση να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη, ως πρόσχημα. Η περιβαλλοντική πολιτική έχει τεράστια σημασία και αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να, να προωθήσουμε και να εγκρίνουμε αυτό το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Περέρο στο συγγνώμη που σα διακόψα λίγο προώρα. Περνάμε στο Catch the Eye και δίνουμε το λόγο πρώτα στην κυρία Θενάσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με χαρά ακούμε ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον θα είναι στη διάθεσή μας στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Πολλά μένουν να γίνουν για το περιβάλλον. Το περιβάλλον πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε άλλη πολιτική, συμπεριλαμβανομένων και των διαρθρωτικών πολιτικών. Χρειαζόμαστε συνεπείς πολιτικές και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οράματός μας για το περιβάλλον. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ουσιαστική υλοποίηση της νομοθεσίας που θα εγκριθεί και επίσης δείκτες περιβαλλοντικούς που θα αντιστοιχίζονται με την υφισταμένη πραγματικότητα. Διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, πολιτική βούληση και κατάλληλη χρηματοδότηση είναι άλλα ε, πράγματα που χρειαζόμαστε. Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 για τη βιοπικιλότητα πρέπει εξάπατος να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα δράσεως για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Αντωνέσκου, λέει ο Πρόεδρος και τώρα ο κύριος Χρούτε. Πρόεδρε, σημαντικό θα είναι στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης να έχουμε ουσιαστική αποτελεσματικότητα, όπως ακριβώς συζητούμε και όπως ασφαλώς θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, όπως έχουμε εγκρίνει άλλωστε στην Επιτροπή μας. Η διάσκεψη για το 2020 θα είναι, πιστεύω, ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έχω πολλές ελπίδες να αυτήν στη διάσκεψη των Υπουργών και ελπίζω ότι μπορούμε να ε, ορίσουμε και ε, προοπτικές από τη διεθνή ε, διάσταση και από το Ρίο συγκεκριμένα μέσα από αυτή. Ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η παραγωγή δηλαδή αυτοκινήτου που θα πρέπει να παρακολουθείται ως προς επιπτώσεις του περιβάλλον από την πρώτη στιγμή μέχρι την ε, έξοδο του οχήματος από το εργοστάσιο. Όλα αυτά για να έχουμε μια ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία του 7ου προγράμματος δράσεως. Ευχαριστώ και η κυρία Μαγκίνες τώρα πάντα στο, στη δικασία Καρστιάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στη συζήτηση, πιστεύω, είναι η σύγκρουση μεταξύ των μακροπρόθεσμων στόχων και των βραχυπρόθεσμων ανησυχιών των πολιτών μας. Όταν λοιπόν μιλούμε για αεφόρο παραγωγή και κατανάλωση, ε, δεν ε, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αηφορία, στο τι εννοούμε ως αηφόρο. Όταν έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, το ζήτημα της ε, αηφορίας δεν συζητείται ως τμήμα του προβληματισμού για την ανεργία. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί είμαι βέβαιη ότι και ε, θέσεις εργασίας ε, θα ενισχυθούν, θα αυξηθούν εφόσον εντάξουμε την αηφορία στον δημόσιο διάλογο και επίσης πιστεύω ότι η πρόταση για την ενσωμάτωση της καθαρότητας των υδάτων και της χρήσης περιζακνιοκτώνων στην προοπτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντική γραφειοκρατική επιβάρυνση. Η κυρία Μαγκίνε, πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαγκίνε. Και έτσι ολοκληρώνεται το Καρστιά για να δώσω το λόγο στον κύριο Ποτόσον, τον Επίτροπο. Thank you. And Ευχαριστώ σα ευχαριστώ όλου για την υποστήριξή σα. Καταρχά θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Για μένα το να τεθεί, το, να υπάρξει ή να μην υπάρξει ένα έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δεν ετέθη ποτέ σαν πρόβλημα, σαν δίλημα. Απλά υπήρχαν ε, κάποιες χώρες οι οποίες ε, θα έπρεπε να, ε, να να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα από το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο και ακόμα και αν υπήρξε ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στο έκτο και στο έβδομο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας ακούμε προσεκτικά και δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία εσείς ζητάτε. Φέτος, σαν παράδειγμα, θα πάρετε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τους υδάτινους πόρους, για τα ορυκτά καύσιμα κτλ. Και τα τελευταία δύο χρόνια θέματα που αφορούν την βιοπικιλότητα, την αποτελεσματικότητα των πόρων κτλ. είναι θέματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απαιτείται όμως να υπάρξει ένα συνεκτικότερο πλαίσιο και πάνω σε αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Δεύτερον να πω ότι έχουμε αρχίσει να πλησιάσουμε σε ένα επίπεδο κοινής κατανόησης των στόχων του εβδόμου προγράμματος, ιδιαίτερα τώρα στο τέλος της εβδομάδας. Στην αρχή της εβδομάδας ε, είχαν ξεκινήσει συζητήσεις και στην Ίγκο και στην Δανία στα πλαίσια της Προεδρίας και τώρα ε, μετά από, μια, από μέρες βλέπω ότι υπάρχει μια σύγκληση για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τι θα πρέπει να αντιμετωπίζει κτλ. Η διαβούλευση η δημόσια είναι ανοιχτή μέχρι τον μήνα Μάιο και περιμένουμε και από εκεί πολλές καλές ιδέες. Να σχολιάσω αυτό το δίλημα λίγο το οποίο μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και την μη πράσινη ανάπτυξη. Ε, το θέμα είναι ότι δεν θα συζητούσαμε για την πράσινη ανάπτυξη αν η άλλου είδους ανάπτυξη δεν ήταν προβληματική και δεν είχε δείξει τα όρια της στον τομέα, τον αναπτυξιακό. Αυτό είναι το βασικό και πολλοί θα πρέπει να το κατανοήσουν. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας λοιπόν τα στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή μας περιορίζουν να μοιραστούμε σωστά τους φυσικούς πόρους όπως ε, τους υδάτινους πόρους, τους ωκεανούς κτλ τότε στην ουσία θα αποκλείσουμε μόνοι μας τις δυνατότητές μας και τις ευκαιρίες μας στο μέλλον. Ένα παράδειγμα, αν συνεχίσουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα, τότε το 2030 που δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, θα χρειαστούμε 40% περισσότερους υδάτινους πόρους από ό,τι έχουμε σήμερα στον κόσμο. Δεν πάει πουθενά λοιπόν αυτή η λογική, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να γίνει δεκτό. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε και σε δείκτες πέραν του ΑΕΠ. Γιατί όχι. Γιατί πράγματι αυτό το οποίο δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει δεν μπορεί να το λάβει και υπόψη του στην πολιτική του και στις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτούς τους άλλους δείκτες. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι διαφορετική από αυτήν που αντιμετωπίζαμε πριν 10 χρόνια στα πλαίσια του έκτου προγράμματος πλαισίου. Έχουμε πολύ περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις διαθέσιμες. Από την άλλη θα πρέπει να κατανοήσουμε και κάποιες νέες προκλήσεις και κάποια προβλήματα τα οποία είναι περισσότερο προφανή σήμερα από ό,τι στο παρελθόν και πρέπει όλα αυτά να ανταλάβουμε υπόψη μας και να τα εντάξουμε στο 7ο πρόγραμμα. Είναι σαφές ότι βιοπικιλότητα, κλίμα, φυσική πόρη είναι οι βασικοί μας άξονες δράσης. Απ' την άλλη όμως δεν θα πρέπει εμείς να επικαλύπτουμε τα μηνύματά μας με αντίστοιχα παρόμοια. Θα πρέπει να δημιουργούμε συνθέσεις, να συγκεντρώνουμε σωστά την προσοχή μας σε να δημιουργούμε οράματα. Ε, μας ε, είπατε ότι θα πρέπει να δώσουμε προσοχή ιδιαίτερη στα χημικά, στην ποιότητα του αέρα, στις αστικές περιοχές κτλ. κτλ. Όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά βασικός μας στόχος είναι διτός. Πρώτον, η εφαρμογή των υπαρχουσών διαστάσεων και αυτών τα οποία ήδη έχουμε αποφασίσει. Γιατί εκεί έχουμε καθυστερήσει και δεν θα έχουμε κάνει τίποτα για την φύση εφόσον τα θέματα πάνω στα οποία έχουμε πάρει αποφάσεις δεν εφαρμόζονται. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν συνομοθέτης θα πρέπει να ενδιαφερθεί και αυτό γιατί τα πράγματα τα οποία αποφασίζεται θα πρέπει να εφαρμόζονται κιόλας. Και ο δεύτερος άξονας ε, είναι η ολοκλήρωση, η συνοχή, την ονομάζουν ορισμένοι, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όλες οι πολιτικές μας να λαμβάνουν υπόψη ότι ζούμε στα πλαίσια ενός σχεδόν διαδραστικού κόσμου πλέον και είμαστε αλληλοεξαρτώμενοι. Στα πλαίσια της επόμενης δημοσιονομικής πρότασης προφανώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και να δώσουμε σωστή αρκετή προσοχή θα έλεγα στα θέματα του περιβάλλοντος. Λοιπόν γενικά δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ το Γιολάινεν. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Ευχαριστώ κύριε Ποτρότσινγκ και τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα λάβει το λόγο για άλλη μια φορά. Το λόγο κύριος Λάινεν εισηγητής για δύο λεπτά. Η συζήτηση απέδειξε ότι υπάρχει συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα έβδομο πρόγραμμα δράσεω και θα ήθελα να ευχαριστήσω του σκιώδει ηγητέ για την υποστήριξη που προσέφεραν και τη συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ποτόσνη και την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν ήταν δεδομένο εκ πρώτη όψου ότι ο καθένα θα ήθελε να προχωρήσουμε σε ένα έβδομο πρόγραμμα δράσεω. Τουλάχιστον αυτό απέδειχθηκε. Τώρα έρχεται η όρια τη συζήτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πόσο χρήσιμο, αν όχι απαραίτητο, θα ήταν ένα

για το περιβάλλον. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, προκαλέσουμε τους υπουργού Οικονομίας και Περιβάλλοντος ε, και πρέπει να απευθύνουμε μία έκκληση για την ε, περιβαλλοντοποίηση, την, το πρασίνισμα δηλαδή της οικονομικής πολιτικής και της ε, πολιτικής εθνικής οικονομίας. Δεν αρκεί δηλαδή μέσα από το περιβάλλον μόνο να επιδιώκουμε τους στόχους μας. Στρατηγική για το περιβάλλον σημαίνει ταυτόχρονα και δημοσιονομική στρατηγική και στη μεσοπρόθεσμη, ε, στο μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικό στρατη... Ε, προγραμματισμό που θα συζητήσουμε θα πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο ε, τα ποσά τα οποία ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ως ιδιαίτερα αφιερωμένα στο περιβάλλον αλλά πολύ περισσότερα και δεν μπορεί η δράση μας να είναι κατά 80% εις βάρος του περιβάλλοντος και να διαθέτουμε 20% των κονδυλίων συνολικά για να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τη ζημιά που έχει γίνει. Κύριε Επίτροπε, περιμένουμε πολύ περισσότερα και καθώς περνάμε από τη διαδικασία της συναπόφασης θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένη η δράση μας. Περιμένουμε να δούμε τις, προτάσεις σας, ε, τις τελικές προτάσεις ε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται η συζήτηση ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα στις 12 και μέχρι τις 12 διακόπτουμε τη συνεδρίαση.